<laughs> Okay, friends, can I suggest that we... Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Ήδη έχουμε καθυστερήσει 15 λεπτά σε σχέση με το πρόγραμμά μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ, ας περάσουμε αμέσως στο επόμενο σημείο που έχουμε στην εμερήσια διάταξη, που είναι το σχέδιο έκθεσης για το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014 με 2020. Θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στον εισηγητή, τον κύριο Όλε Κρίστενσεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην έκθεση αυτή πρωτοβουλίας. Έχω πάρει πολλά mail, γράμματα από συνδικάτα, από εργοδότε κλπ. Η ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το στρατηγικό αυτό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014 και 2020 τελικά τον Ιούνιο πέρυσι εγκρίθηκε. Έχω δύο γενικές σκέψεις πρώτα απ' όλα για το στρατηγικό αυτό πλαίσιο που αντικατοπτρίζονται και στο σχέδιο εκθεσής μου. Νομίζω λοιπόν το στρατηγικό πλαίσιο πολύ καλά κάνει που αναφέρει τις κύριες προκλήσεις της Ευρώπης σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Υπάρχουν νέα αναδυόμενοι κίνδυνοι και ασθένειες που συνδέονται με την εργασία επίσης. Η εφαρμογή είναι πολύ σημαντικό και εμπίπτει στα πλαίσια της εθνικής στρατηγικής, όπως επίσης και τα στατιστικά δεδομένα που έχουν να κάνουν με την γύρανση του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα συγκεκριμένες δράσεις, το στρατηγικό πλαίσιο δεν είναι αρκετό. Οι εργοδότες, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα που απαιτούν συγκεκριμένες δράσεις. Συνεπώς, η έκθεσή μου προσπαθεί να προτείνει κάποιες λύσεις και ελπίζω και προσδοκώ επίσης ότι εμείς ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε πάνω σε μια ρεαλιστική θέση και έτσι να συνεισφέρουμε σε μελλοντικέ νομοθετικές πρωτοβουλίες όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Με άλλα λόγια, χρειάζονται πιο συγκεκριμένα μέτρα και νομοθετικά μέτρα που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει κατ' εμέ το στρατηγικό πλαίσιο. Πρώτον είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε υψηλότατο επίπεδο προστασίας όταν πρόκειται για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης στην οποία δουλεύουν. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει και να εφαρμόζει συγκεκριμένους στόχους ποσοτικούς ε, που θα τους μειώσει όσον αφορά τους κινδύνους και τις ασθένειες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, το προηγούμενο στρατηγικό πλαίσιο. Οι εθνικές στρατηγικές τώρα. Αυτό που ακούμε από τους κοινωνικούς εταίρους και τους εργοδότες είναι ότι η εισαγωγή εθνικών στρατηγικών είναι κάτι που απορρέει από την παλιότερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ήταν επιτυχισμένη, αλλά πρέπει να είναι περισσότερο διάφανη και να επιτρέπει και τη συμμετοχή των συνδικάτων και άλλων εταίρων. Πρέπει επίσης να έχουμε και εκθέσεις και αναφορές όσον αφορά την πρόοδο που επιτυχάνεται. Πρέπει να υπάρχουν ίσες, ίδιες μάλλον και οι κανόνες εδώ έχουν τεράστια σημασία γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες που εγκρίνουμε θα είναι προ όφελο των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η αποτελεσματική επίσης εφαρμογή και επιβολή των μέτρων είναι ζωτική σημασία για να πετύχουμε μια κατάσταση που θα προστατεύει εξίσου όλου. Η συμμόρφωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τώρα. Η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη πρέπει να φροντίσουν για τη συμμόρφωση αυτή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να εκπονήσουν συγκεκριμένα εργαλεία και κατευθυντήριε γραμμέ για να βοηθήσουν στη συμμόρφωση αυτή. Η κοινωνική εταίροι τώρα και εκπρόσωποι των εργαζομένων. Η αξιολόγηση, όπως επίσης και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και ιδιαίτερα των εργαζομένων και των εκπροσώπων του σε επίπεδο επιχείρηση είναι ζωτική σημασία για να διευκολύνει την αποτελεσματική συμμόρφωση και επιβολή των μέτρων επιθεωρήσεις, επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και να υπάρχουν και κατάλληλοι πόροι για να έχουμε και αρκετούς επιθεωρητές να κάνουν τις επιθεωρήσεις αυτές. Οι χώρες μέλη πρέπει να ακολουθήσουν τις συστάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που μιλάει για έναν επιθεωρητή ανά 10.000 εργαζόμενους. Όσον αφορά τώρα τις ασθένειες που έχουν να κάνουν με τους χώρους εργασίας, όντως υπάρχουν νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι και ασθένειες που συνδέονται με την εργασία. Και αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί. Οι, μικρομεσές, ε, συγνώμη, οι χώρες μέλη, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η απουσία από τους χώρους εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τις μέχρι τώρα προτάσεις μέσα σε μια συνολική οδηγία ώστε να προστατεύονται οι εργαζόμενοι από εργονομικούς κινδύνους. Οι εργοδότες θα πρέπει να επεκτείνουν τα ευρωσεφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φροντίσουν για ρυθμιστικά πλαίσια ώστε να εφαρμόζουν τις ευρωπαϊκές ε, συστάσεις. Είτε πρόκειται για φόνες που χρησιμοποιούν εργαζόμενοι είτε για άλλους παράγοντες που προκαλούν διαταραχές. Πρέπει επίσης να υπάρξουν και περισσότερα δεσμευτικά επίπεδα ε, έκθεσης σε καρκινογενείς παράγοντες ή μεταλλαξιογόνους. Χρειάζεται στενή συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και ένα σύστημα το οποίο να επιτρέπει την πρόσβαση στα όρια έκθεσης που να εξηγούνται απλά και κατανοητά. Υπάρχουν επίσης και ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στους χώρους εργασίας. Εδώ αυτό που χρειαζόμαστε είναι καλύτερη συλλογή στοιχείων και έλεγχο. Άλλοι τομείς που μας απασχολούν είναι το θέμα της έκθεσης των αμίαντο και η νανοτεχνολογία. Χρειάζονται περισσότερα και πιο αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα. Αυτό είναι κάτι που επανέρχεται κάθε φορά που συζητάμε με τους κοινωνικούς ε, εταίρους. Αξιόπιτα στοιχεία μας επιτρέπουν να θέσουμε στόχους και να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές στις χώρες μέλη. Δεν μπορέσαμε βέβαια να συμπεριλάβουμε όλες τις προτεραιότητες στην ε, έκθεση αυτή εξαιτίας του περιορισμού που έχουμε για το περιεχόμενο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι με τροπολογίες θα εμπλουτίσουμε την έκθεση αυτή, όπως επίσης θα εμπλουτιστεί και από τις νομοδοτήσεις της Επιτροπής για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Και θα σταματήσω εδώ, προκειμένου να ακούσουμε και τους προσκεκριμένους μας και τους σκιώδες εισηγητές. Προσβλέπω στη συνέχεια της συνεργασίας μου μαζί σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή και θα ήθελα να δώσω κατευθείαν το λόγο τώρα στους προσκεκλημένους μας. Ο πρώτος εξ αυτών, λοιπόν, είναι ο επικεφαλής, η επικεφαλής η κυρία Γκρίστα του ΟΣΚΕ. Έχει το λόγο λοιπόν, του Όσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Κρίστενσε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου. Μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα και χαίρομαι που μπορώ να συμβάλλω στο θέμα του ευρωπαϊκού στρατηγικού πλαισίου, στο θέμα της ε, ασφάλειας των χώρων και θα παρουσιάσω το ρόλο της, ε, του Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές, αλλά θα ήθελα να τονίσω επίσης ασφαλώς ότι με χαρά θα συμβάλλουμε στο πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται στην παρούσα φάση και θα ήθελα ο συναδελφός μας να παρουσιάσει ένα από τα βασικά μας προγράμματα, μία μελέτη για να παρουσιαστούν και τα σχετικά στοιχεία. Ξεκίνησε σήμερα στο Κοινοβούλιο η παρουσίασή του, θα αποτελέσει βασική πηγή δεδομένων και για χρήση στο στρατηγικό πλαίσιο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με μια ιστορική αναδρομή σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και την υπηρεσία μας. Τα θέματα αυτά πάντα εντοπίζονταν ως μια ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι καινούργοι αλλά και οι πιο παλιοί κίνδυνοι στον χώρο της εργασίας. Από το 2002 ήδη η στρατηγική για το πλαίσιο του 2002-2006 τόνισε ότι οι νέοι και οι παλιοί κίνδυνοι που προκαλούνται από τις τεχνικές καινοτομίες ή από την κοινωνική εξέλιξη θα πρέπει να εντοπίζονται γιατί αυτό αποτελεί κατεμπίγουσα ανάγκη καθώς και ο έλεγχος τους και ότι αυτό σημαίνει καταρχάς παρατήρηση των ίδιων των κινδύνων βάσει μιας συστηματικής συλλογής τέτοιων επιστημονικών στοιχείων και γνωμοδοτήσεων. Από τότε λοιπόν ο ρόλος μας ήταν ουσιώδης στην περίοδο 2002 έως 2006 οι στρατηγικές μας ε, έθεσαν ε, την, ε, επικεντρώθηκαν στη δημιουργία ενός παρατηρίου για την εκπλήρωση των καθήκοντων αυτών και αυτό διευκρινίστηκε στην περίοδο 2006 έως 2012 και εκεί τονίστηκε η σημασία πρόβλεψης των κινδύνων και στήθηκε από το παρατηρητήριο να λάβει μια σειρά πρωτοβουλειών. Τώρα, το 2014 ξεκίνησε το στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασία μέχρι την ε, περίοδο του 2020 και υποστηρίζονται περαιτέρω τα ευρήματα του παρατηρητηρίου. Και εδώ τονίζουμε ότι στο στρατηγικό πλαίσιο αυτό θεωρούμαστε ένας από τους βασικούς παράγοντες στο στρατηγικό λοιπόν πλαίσιο εντοπίζονται, όπως είπε και ο κύριος Κρίστενσεν, οι βασικές προκλήσεις. Και τι οι στρατηγικοί στόχοι μέχρι το έτος 2020. Όπως σας είπα λοιπόν η όσα ήδη διατραματίζει σημαντικό ρόλο για την εφαρμογή της ήδη φυσάμενης στρατηγικής για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και σε ό,τι αφορά την εξωτερική αξιολόγηση της στρατηγικής. Στο νέο στρατηγικό λοιπόν πλαίσιο, η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τις εθνικές ε, πολιτικές για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Εδώ συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναπτύσσουμε νέα εργαλεία παρακολούθησης αλλά και παρουσίασης των εθνικών στρατηγικών για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί είναι η συμμόρφωση με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την υγεία των τόπο Και επίσης ε, ξέρετε ότι εκτελούμε ένα τεράστιο project έργο που μας ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα παρουσιάσουμε τα σχετικά ευρήματα στα τέλη του έτους σε μια σχετική μερίδα και στις αρχές του 2016 θα παρουσιάσουμε τελικά πορίσματα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις τελικές συστάσεις. Ένας άλλος τομέας είναι η αναδυόμενοι νέοι κίνδυνοι και αυτό συνδέεται με την μελέτη την οποία θα σας παρουσιάσουμε λίγαν συντόμως. Ε, μια άλλη σημαντική πτυχή είναι η πρόληψη των ε, ασθενειών που προκύπτουν από το, την εργασία και η πρόληψη πρακτικής βοήθειας, η παροχή πρακτικής βοήθειας σε μικρές ε, επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα λοιπόν για αυτές τις πολύ μικρές επιχειρήσεις έχει αναπτυχθεί ένα εργαλείο online, το OIRA, για την αξιολόγηση κινδύνων για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και πάλι στο στρατηγικό πλαίσιο ζητείτε να αναπτύξουμε ιδιαίτερα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις πρακτικά εργαλεία που θα βοηθήσουν τις εταιρείε αυτές να εφαρμόσουν τα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Και αυτό αποτελεί λοιπόν το σύνδεσμο με την επόμενη παρουσίαση και εδώ θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο William Κόμπορν που θα παρουσιάσει τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την μελέτη αυτή. Σα ευχαριστώ, Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητοί βουλευτές που μα δίνετε το λόγο να παρουσιάσουμε την ε, μελέτη αυτή. Είναι μια συναρπαστική νέα πρωτοβουλία, μια νέα ομάδα δεδομένων που σίγουρα θα είναι ωφέλιμη για τις συζητήσει σα. Η Ευρωπαϊκή Μελέτη για του νέου Αναδυόμενου Κινδύνου είναι μια μελέτη που έγινε για πρώτη φορά το 2009. Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση και τελείωσε η συλλογή στοιχείων πέρσι και παρουσίασαν τα πρώτα πορίσματα στι αρχέ του φετινού έτου. Όπω είπε και η διευθυντριά μου, σήμερα είναι η μέρα που ξεκινάμε την πρώτη ε, σύνοψη των βασικών πορισμάτων και με χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο. Στην παρουσίαση που θα είναι πολύ σύντομη, θα ήθελα να σα δώσω μια σύντομη επισκόπηση τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, να επικεντρωθώ στα πολύ βασικά πορίσματα και να σχολιάσω εν συντομία το πώς αξιολογούμε και αξιοποιούμε τις, ε, τα δεδομένα αυτά στις μελλοντικέ μας δραστηριότητε. Για να απαντήσω καταρχάς ένα σημαντικό ερώτημα. Για να δούμε τις διαφάνειες. Γιατί χρειαζόμαστε άλλη μία μελέτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν ε, μία σειρά πηγών δεδομένων, τις οποίες θα γνωρίζετε πολύ εξημών. Έχουμε μελέτες που γίνονται με το ερωτικό δυναμικό διαφόρων χωρών. Έχουμε και τις μελέτες της Eurostat με το τμήμα ad hoc που αφορά τις ασθένειες και τα ατυχήματα. Έχουμε επίσης ε, την Eurofound ε, που είναι αδελφή υπηρεσία και κάνει επίσης παρόμοιες μελέτες κοιτώντα τα διοικητικά στοιχεία από την Eurostat για τα ατυχήματα στο χώρο εργασίας έχουμε και τις στατιστικές για τις ε, ασθένειες στον χωροεργασία. Το Το πλεονέκτημα της ε, ευρωπαϊκής αυτής βάσης δεδομένων είναι ότι μπορούμε να κάνουμε μια συγκριτική ανάλυση και να διδαχτούμε από τις διαφορές που υπάρχουν βάσει των δεδομένων και από την κατάσταση που υπάρχει στα διάφορα κρατημέλη. Ε, κατά πάσα πιθανότητα αυτό οφείλεται στις διαφορετικές πολιτικές που ακολουθούνται. Έχω κάποιο πρόβλημα με διαφανίες μου δεν ακολουθούν τη σειρά που ήθελα. Μάλιστα. Ας συνεχίσω λοιπόν να αναφέρω τι μελέτες αυτές που έχουμε για το εργατικό δυναμικό και τα δυτικά στοιχεία μας δίνουν μια καλή εικόνα σε όλη την Ευρώπη για τους τραυματισμούς και τις ανησυχίες που υπάρχουν στο εργατικό δυναμικό. Λιγότερο όμω, καλύτερη, καλή εικόνα για τι εργασιακέ ασθένειε. Έχουμε πάρα πολύ λίγε πληροφορίε που συνδέουν τι πρωτοβουλίε τη πολιτική με αυτά που συμβαίνουν στον χώρο εργασία. Και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα σύνδεση μεταξύ τη πρωτοβουλία για την πολιτική και του αποτελέσματο. Σε Ιέσνερ, λοιπόν εστιάζεται στην μελέτη του τι ακριβώ γίνεται ω προληπτική δράση στου χώρου εργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύπτονται 36 χώρες, 28 ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Αλβανία, η πρώην Ιγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Ισλανδία, η Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία. Η Ελβετία θεώρησε ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία για να πληρώσει και το βασίλεια Βασίλειο, Ισπανία και η Σλοβενία πλήρωσαν από τα κονδύλια τους για να, αυξήσει, να αυξήσουν τη δεγματοληψία και να αντικαταστήσουν έτσι η εθνική μελέτη περίπου 50.000 υπηρεσίες. Πολύ δηλαδή μεγάλος αριθμός υπηρεσιών κάλυψαμε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στους δύσκολα προσβάσιμους, όπως η γεωργία και η αλληλεία, που είναι πολύ σημαντική τομής όμως για, σε διαφορά αφορά το σκέλος της πρόληψης. Και το πιο σημαντικό, ανταποκρινόμενοι στις ε, απαιτήσει των ε, φορέων, μειώσαμε την δειγματοληψία σε επιχειρήσεις ε, σε ό,τι αφορά τι μικρές επιχειρήσεις με λιγότερο από πέντε απασχολούμενους ε, μάλλον πήραμε δειγματοληπτικό δείγμα και από μικρές μικρές επιχειρήσεις ε, με λιγότερο από πέντε απασχολ... Ε, υπαλλήλους. Δύσκολο αλλά απαραίτητο. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ποιους, με ποιου μιλήσαμε, ποιους ρωτήσαμε σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασία τους. Επικεντρωθήκαμε λοιπόν στα άτομα τα οποία γνωρίζουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τι γίνεται στην πράξη για την οργάνωση της υγείας και της ασφάλειας και βρήκαμε λοιπόν τον εξή ορισμό βάσει των εμπειριών της πρώτης έρευνας και στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους οδηγηθήκαμε σε αυτή την ενέργεια. Έχουμε διάφορες απαντήσεις. Έχουμε διάφορα άτομα λοιπόν τα οποία ρωτήσαμε στις στερήσεις, στους διευθυντές, στους ιδιοκτήτες και στις μικρές επιχειρήσεις από ό,τι φαντάζεστε. Όσο πιο μικρή είναι η επιχείρηση, τόσο λιγότερο πιθανό είναι το άτομο αυτό το οποίο είναι υπεύθυνο για θέματα υγείας και ασφάλειας. Όσο πιο μεγάλη είναι η εταιρεία, τόσο πιο πιθανό είναι να υπάρχει κάποιο υπεύθυνο για θέματα ασφάλεια που απασχολείται από τη διευθυνσή. Αλλά σε όλα τα μεγέθη 20% των ερωτηθέντων ήταν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων για θέματα υγείας και ασφάλειας. Αυτοί λοιπόν προβάλλονται ως άτομα υπεύθυνα για να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Αυτό τονίζει ότι οι διατάξεις στον χώρο εργασίας δεν έχουν οργανωθεί με τον βέλτιστο τρόπο, όπω υπονοείται σε κάποιε περιπτώσει στη συζήτηση για την πολιτική. Ποια είναι τα αποτελέσματα λοιπόν, τα βασικά απορίσματα, ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντε που αποτελούν. Ε, που απειλούν την υγεία και την ασφάλεια. Βλέπετε από τα παραδείγματα ότι καταρχάς αντιμετωπίζουμε δύσκολους ε, ε, πελάτες, ασθενείς ή μαθητές. Η πίεση, η χρονική η ανεπαρκής επικοινωνία των στόχων και των αποτελεσμάτων. Αυτό καταδεικνύει ότι είναι ψυχοσωματική, ψυχοκοινωνική η κίνδυνη ως επιτοπλίστων. Ωραία. Μια και δουλεύουμε διαφάνειες, κοιτάξτε τα αντιτύπα που έχετε και πώς αυτή η ψυχοκοινωνικοί παράγοντε κινδύνου είναι βασική. Ύστερα, οι διαταραχές ε, μειοσκελετικές ε, λόγω επαναληπτικών κινήσεων ε, καθιστικής ζωής και εργασιακής ζωής δηλαδή. Και αυτά τονίζονται στο στρατηγικό πλαίσιο. Πώς λοιπόν αυτοί οι παράγοντες κινδύνου αντιμετωπίζονται στο χώρο εργασίας. Εδώ γίνεται καταρχάς μια μελέτη αντικτύπου και αξιολόγηση κινδύνου. Ο εργοδότης ως υπεύθυνο ελέγχου της διαδικασίας ε, στην εργασία ξέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτοί οι κίνδυνοι και είδαμε μεγάλες αποκλήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Μεγάλη ποσοστό αξιολόγηση κινδύνου στην Ιταλία, 85% μέχρι 35% στο Λουξεμβούργο αντίστοιχη αξιολόγηση κινδύνου. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι δεν μιλάμε για συμμόρφωση, για συμμόρφωση με τις νομικές μετάξεις, μιλάμε για την αντίληψη των εταιριών για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Μιλάμε για μια εκτίμηση. Και οι, οι επιχειρήσει ε, παροχή υπηρεσιών έχουν λιγότερε πιθανότητε σε ε, διεξαγωγή τέτοια αξιολόγηση κινδύνου, όπω αντίστοιχα και οι μικρέ επιχειρήσει έχουν μικρότερη πιθανότητα διεξαγωγής αξιολόγησης κινδύνου. Γιατί λοιπόν κάποιες εταιρείε έχουν ε, τόσο μεγάλη δέσμευση για την ε, πρόληψη τέτοιων κινδύνων. Συνήθως μας θέλανε για να πληρούν τις νομικές τάξει. Και σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της επιθεώρησης εργασίας. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η νομοθεσία και η εφαρμογή της νομοθεσίας και ο έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας. Δεύτερος λόγος για την έλλειψη δράψης είναι οι προσδοκίες των ε, ε, υπαλλήλων από την διοίκηση. Και αυτό καταδεικνύει ότι μία επιχείρηση όπου υπάρχουν τις προσδοκίες έχει 10 πλάσιες πιθανότητες να λάβει προλεπτικά μέτρα. Και εδώ αναφέρεται πάρα πολύ στα νέα κρατημέλη, ιδιαίτερα σε σχέση με τα παλιά κρατημέλη, το θέμα της φήμης της εταιρεία. Γιατί λοιπόν οι εταιρείε ε, λαμβάνουν δράση, γιατί οι εταιρείε αποφασίζουν αντίστοιχα να μην λάβουν δράση και δεν ε, λαμβάνουν προληπτικά μέτρα. Βλέπουμε ότι τα βασικά προβλήματα είναι οι κίνδυνοι, οι οποίοι είναι ήδη γνωστοί, η αντίληψη για κάποια προβλήματα. Πολύ πιο πολύ σημαντικό παράγοντας σε σχέση με το πόσο βαριά είναι η διαδικασία, πόσο α, βαρύνει βαραίνει η έλλειψη εμπειρογνωμοσύνη. Αλλά όλε οι επιχειρήσει καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν κίνδυνοι ανεξάρτητα από τον τομέα, ανεξάρτητα από τον, ε, το μέγεθο τη επιχειρήση. Όταν ρωτήσαμε για την αξιολόγηση κινδύνου, το 90% μα είπαν ότι η αξιολόγηση κινδύνου είναι η πιο, σωστός, ε, η πιο σωστή μέθοδο αντιμετώπιση των κινδύνων. Στην επόμενη διαφάνεια. Ρωτήσαμε ποια είναι τα εμπόδια σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των θεμάτων υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Για, λόγω τη περι, περιπλοκότητα τη νομοθεσία και εδώ στην Ιταλία, 70% των επιχειρήσεων μα είπαν ότι η περιπλοκότητα τη νομοθεσία αποτελεί τη μέγιστη δυσκολία. Στη Σλοβανία και στην ε, Λιθουανία τα ποσοστά αυτά είναι περίπου 40% και 84% δηλώνει ότι δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα το πόσο περίπλοκη είναι η νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις ε, λειτουργούν με το ίδιο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Βλέπουμε όμως ότι είναι διαφορετικές καταστάσεις στα κράτη-μέλη και αυτό τροποποιεί το πώς αντιλαμβάνονται την νομοθεσία οι επιχειρήσεις. Στην επόμενη διαφάνεια αναρωτιόμαστε οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει έχουν έλλειψη πληροφοριών για την αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνων. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω κάποιους παράγοντε κινδύνων που ανέφερα στην αρχή τη παρουσίαση, σε ό,τι αφορά την ανασφάλεια τη θέση εργασίας, της έλλειψης επιρροή που συνδέεται πιο πολύ με του ψυχοκοινωνικού παράγοντες κινδύνου. Και εδώ οι πιο πολλέ επιχειρήσει δηλώνουν ότι δεν υπάρχει καθοδήγηση και δεν ξέρουν πώ να αναλάβουν προληπτική δράση. Έτσι καταδεικνύεται λοιπόν από τη μελέτη μας ότι εδώ πέρα μπορεί να υπάρξει μεγάλη πρόοδος. Αναρωτιόμαστε επίσης ε, κατά πόσον οι εργάτες μπορούν να συμμετέχουν και να επηρεάσουν το πώς ε, ε, αντιλαμβάνονται και πώς αντιμετωπίζουν τα θέματα υγείας και ασφάλειας. Αν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος ε, των υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι λοιπόν έχουν ένα ρόλο να διαδραματίσουν, αλλά σε πολύ διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με το κρατό μέλο, σε, σε ό,τι αφορά του ψυχοκοινωνικού παράγοντε κινδύνου. Εδώ χρειάζεται, όπω ξέρουμε, μεγάλη συμμετοχή των υπαλλήλων, αν θέλουμε να υπάρχει επιτυχία. Επίση, λόγω τη οδηγία πλαισίου στι μικρέ υπηρεσίε υπάρχουν καν οι εκπρόσωποι των υπαλλήλων και των ε, εργασιακών δυνάμεων. Στην τελευταία διαφάνεια, γιατί δεν έχω και χρόνο, θα ήθελα να σας παρουσιάσω μια εικονική, μια απεικόνηση του τι γίνεται. Και βλέπετε λοιπόν ότι μπορείτε να βρείτε μέσα στην ιστοσελίδα μας ε, με μια οπτική απεικόνηση όλες τις ερωτήσεις που σας ανέφερα, μια μικρή μόνο, ένα μικρό μόνο κλάσμα των ερωτήσεων που διαπραγματευτήκαμε ε, σας ανέφερα εδώ σήμερα για να τα συμπεριλάβετε όλα αυτά στις συζητήσεις σας. Την ιστοσελίδα μας θα τη βρείτε στην τελευταία διαφάνεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που μας μεταδώσατε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τους κοινωνικούς εταίρους. Τους έχουμε μαζί μας σήμερα και θα ήθελα να δώσω το λόγο τον πρόεδρο της ομάδας ασφαλείας και συνθήκων εργασίας του Business Europe. Ο κύριος Τεμέστερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι πιστεύουμε ότι απαιτείται ένα περιβάλλον για τις επιχειρήσεις ασφαλές, όχι μόνο σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας, αλλά και σε επίπεδο συνθήκων εργασίας. Η προστασία των ε, εργαζομένων είναι απαραίτητο για μας στο Business Europe. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που τα πάνε καλά, παίρνουν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και έχουν αρκετά υψηλά επίπεδα συμμετοχής και εμπλοκής των εργαζομένων. Υπάρχουν σημαντικές διαφοράσεις βέβαια ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ανάμεσα στους διάφορους τομείς. Θα ήθελα να μοιραστώ επίσης μαζί σας και κάποιες ανησυχίες που έχω σχετικά με την έκθεση. Καταρχάς, ποιος είναι ο σωστός δρόμος για την ανάληψη της κατάλληλης δράσης. Κατάλληλη δράση όταν λέμε δεν είναι κάτι το οποίο υποχρεωτικά είναι νέα νομοθετικά μέτρα. Εξακολουθούμε εμείς να ελέγχουμε την αξιολόγηση της υπάρχουσας νομοθεσίας και νομίζω ότι η αξιολόγηση των δράσεων που έχουν ε, ήδη ε, αναλυθεί ε, και η σωστή εφαρμογή τους είναι απαραίτητη πριν αποφασίσουμε νέα μέτρα για το μέλλον. Όπως και να έχουν τα πράγματα, η στάση γενικότερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται στην σωστότερη εφαρμογή, τη συμμόρφωση των νομοθετικών ρυθμίσεων εθνικών και κοινοτικών. Όπως είπα, φυσικά σε μια δεύτερη φάση θα δούμε την περαιτέρω νομοθετική ε, ρύθμιση. Ίσως εδώ να δώσω κάποια στοιχεία ανησυχίας που έχουμε γύρω από την πρόταση επιβολής ποσοτικά, ποσοτικών μειώσεων σε κοινοτικό επίπεδο. Νομίζω ότι η δομή του πλαισίου αυτού έχει σαν στόχο να εντοπίσει τις βασικές προκλήσεις χωρίς να περάσουμε σε αυτή τη φάση σε ποσοτικές μειώσεις. Δηλαδή, πρακτικές μηδενικού ατυχήματος όπως ε, τις λέμε, υποστηρίζουμε τέτοιου είδους αντιλήψεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι μεταφράζεται αυτό άμεσα σε ποσοτικό στόχο μηδέν. Ε, τα προγράμματα αυτά μηδενικού ατυχήματος είναι θα έλεγα εφαρμογή μιας συνολικότερης λογικής και πολλαπλών μέτρων μέτρα τα οποία έχουν σαν στόχο το μηδέν, αλλά το θέμα δεν είναι να πετύχουμε το μηδέν απλά, αλλά τι κάνουμε για να φτάσουμε εκεί. Υπήρχε ένας τέτοιος ποσοτικός στόχος και είπαμε επίσης ότι και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες το έχουμε σαν στόχο. Όχι αν πετύχαμε το στόχο, αλλά το τι κάνουμε για να πετύχουμε το στόχο, αυτό έχει σημασία. Η αξιολόγηση των κινδύνων, τώρα η εκτίμηση των κινδύνων έχει σημασία σε σχέση με την αξιολόγηση των κινδύνων. Να πούμε ότι είναι μια διαδικασία η οποία έχει σαν στόχο, έναν στόχο υψηλό. Ο υψηλός αυτός στόχος είναι πρώτον η διαμόρφωση των κατάλληλων, η μορφοποίηση καλύτερα των κατάλληλων μέτρων προστασίας των εργαζομένων και δεύτερον η σωστή εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών. Στόχος δεν είναι να αξιολογήσουμε θεωρητικά τον κίνδυνο, αλλά να χρησιμοποιήσουμε την αξιολόγηση του κινδύνου για να βρούμε μέτρα για να τον αποφύγουμε. Εκεί θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας και όχι στο ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει κάθε μία να έχει ένα συγκεκριμένο έγγραφο για την αποφυγή του κινδύνου, αλλά οι διαδικασίες αυτές πρέπει να είναι εφαρμοστές. Ένα άλλο στοιχείο αφορά τα προβλήματα υγείας, τα μειοσκελετικά. Είναι ένα σημαντικό θέμα ε, το θέμα είναι βέβαια τι δράση μπορούμε να αναλάβουμε. Δεν νομίζω ότι ε, η νομοθετική δράση είναι κάτι το οποίο θα λύσει αποκλειστικά τα χέρια μας. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από τους παράγοντες κινδύνου έχουν ήδη εντοπιστεί και σε εθνικό επίπεδο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Δεν είναι νομοθετικό το πρόβλημα εδώ. Δεν χρειάζεται να συζητήσω το γεγονός ότι η αντιμετώπιση ε, του προβλήματος αυτού είναι ε, πολυπαραγοντική, αλλά απαιτείται η σωστή ισορροπία μέτρων. Τώρα, για κάποιες ασθένειες που προκαλούνται από την απασχόληση έχουμε ανάγκη από περαιτέρω αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα. Ποτέ δεν έχουμε κάτι τέτοιο και ποτέ δεν θα το αποκτήσουμε φοβάμαι. Πόσα χρόνια συλλέγουμε στοιχεία και στατιστικές, στατιστικές για ατυχήματα. Έχουμε χιλιάδες δεδομένα για επιχειρήσεις, έχουμε και την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα, αλλά δεν είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα αυτά. Οι Φιλανδοί συναδελφοί έκαναν κάποιες συγκρίσεις για τις βαλτικές και σκανδιναβικές χώρες και ούτε εκεί δεν μπορούν να κάνουν τις συγκρίσεις και μιλάμε για γενικής φύσης δεδομένα. Τα δεδομένα που είναι χρήσιμα είναι τα μικροδεδομένα. Μια επιχείρηση γνωρίζει και ελέγχει το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της και λαμβάνει τις απαιτούμενες δράσεις. Αν έχει κανείς συνολικά, ε, ε, ε, συνολικές συνθέσεις τέτοιων δεδομένων και σε εθνικό επίπεδο και σε τομεακό επίπεδο δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Και δεν θα βοηθήσει εν πάση περιπτώσει να προχωρήσουμε. Λοιπόν, τους ζητάμε να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στην ποιότητα των δεδομένων και τα δεδομένα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα ακριβώς στην κατάλληλη μορφή. Το θέμα της ασφάλειας στο χώρο εργασίας ε, είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία αλλά δεν αναφέρεται σε θέματα που άπτονται κοινωνικών όπως λέμε κινδύνων. Το θέμα είναι να βρούμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στις ικανότητες και τις προσδοκίες του εργαζομένου και στην αποστολή την οποία έχει και εδώ τίθεται και το θέμα της στήριξης του εργαζομένου από τους συναδέλφους του και από την εργοδοσία. Αυτό θα πρέπει να ισχύει για το σύνολο της εργασιακής ζωής ενός ε, ε, υπαλλήλου. Το θέμα δεν είναι μόνο ε, το σύνθημα καλύτερη δουλειά, καλύτερες θέσεις δουλειάς. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στη βελτίωση των συνθήκων εργασίας αλλά και στην ύπαρξη ανθρώπων που είναι σε σχέση να σχεδιάσουν τις σωστές σχέσεις εργασίας, να ανοιχνεύσουν το πού υπάρχουν σωστά παραδείγματα και να δούνε αν οι θέσεις αυτές απασχόλησης καλύπτουν τις απαιτούμενες ανάγκες, είναι θέσεις ανθεκτικές, είναι θέσεις ε, οι οποίες επιτρέπουν στον εργαζόμενο να μην κάνει τα ίδια και τα ίδια σε όλη του τη ζωή, γιατί αυτό θα τον οδηγήσει σε μια έλλειψη ισορροπία σε κάποια φάση. Το θέμα είναι να ισορροπήσουμε σωστά τις ικανότητες με το περιεχόμενο της απασχόλησης και εδώ τίθεται και το θέμα της κινητικότητας στην απασχόληση. Πρέπει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν, να έχουν φιλοδοξίες και να συνειδητοποιούν ότι οι επιλογές τις οποίες κάνουν δεν αφορούν μόνο τα εισοδήματά τους αλλά και τα ψυχοκοινωνικά τους χαρακτηριστικά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κέμπα τώρα. Από το UEC. Ερευνητής. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να αρχίσω με ένα γενικό πλαίσιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 έχουμε 10 εκατομμύρια τραυματισμούς πάρα πολλούς θανάτους στους χώρους εργασίας. 200.000 χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που έχουν να κάνουν με την εργασία. Οι τραυματισμοί και οι ασθένειες είναι 3 με 5% του ΑΕΠ. Αυτό λοιπόν Είναι σαφέ ότι χρειάζεται ένα πρόγραμμα δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι σήμερα ζούμε σε ένα κόσμο όπου οι συνθήκε εργασία επιδεινώνονται όχι μόνο εξαιτία τη οικονομική κρίση που οι δαπάνε ε, στον τομέα της υγείας και της ασφάλεια μειώνονται, αλλά και εξαιτία των λάθο αποφάσεων στα διάφορα προγράμματα μειώνεται η νομοθεσία που είχε αναπτυχθεί μέχρι τώρα εξαιτία των κακών συνθηκών που επικρατούν στους χώρους εργασίας και έτσι οδηγούμαστε σε ατυχήματα και σε ασθένειες. Είμαστε επίσης μάρτυρες της κακής επιθεώρησης που γίνεται. Δεν μειώνονται οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, αντίθετα, και αυξάνουν και οι ανισότητες μεταξύ των χωρών μελών αλλά και μέσα στην κάθε χώρα μέλος. Η υπηρεσία μας σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε εκπονήσει διάφορα ψηφίσματα όσον αφορά το λεγόμενο στρατηγικό πλαίσιο σήμερα. Έτσι το ονομάζουμε σήμερα. Εκτιμούμε λοιπόν την έκθεση του κύριου Κρίστενσεν όλος ιδιαίτερος, κυρίως επειδή ζητάει συγκεκριμένες απτές δράσεις. Αυτό που λείπει στο στρατηγικό πλαίσιο σήμερα είναι μετρήσιμοι στόχοι, δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και αξιολόγηση. Ζητούμε επίσης καλύτερη προστασία των εργαζομένων από τα ατυχήματα και τις ασθένειες αντί να μειώνεται η σχετική νομοθεσία ως αντίδραση στην οικονομική κρίση. Οι νομοθετικές προτάσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τους κοινωνικούς εταίρους. Έχουμε τις συμφωνίες για τους κομωτές, ε, που όμως έχουν βλοκαριστεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να παραμείνουν σε επίπεδο οδηγίας για το μέλλον δεν έχουμε και τριμερείς διαλόγους. Αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να στηρίξει τη γνώση όσον αφορά τις επιθεωρήσεις. Δεν έχουμε ούτε κατευθυντήριες γραμμές προς τις χώρες μέλη για να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνεται ε, υπό την εποπτεία της ε, επιθεώρησης του χώρους εργασίας. Ποιες είναι τώρα οι κύριες προτερότητες που πρέπει να συμπεριληφθούν στο τρέχον στρατηγικό πλαίσιο. Τώρα που μετονομάστηκε σε στρατηγική. Θέλουμε δεσμευτικά όρια έκθεσης για να περιοριστούν οι τοξικές ουσίες. Θέλουμε επίσης να βελτιωθεί η υπάρχουσα νομοθεσία όσον αφορά την ε, έκθεση των εργαζομένων σε, καρκοκι... σε καρκινογενείς και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Η σχετική οδηγία δεν υπάρχει ακόμα. Υπάρχουν βέβαια κάποια, κάποιες ρυθμίσεις για τους αντι ενδοκρι... ενδοκρινικούς διαταράκτες, αλλά πρέπει να γίνει ενημέρωση γιατί πολλές φορές τα στοιχεία που έχουμε, τα δεδομένα και οι πληροφορίες στις ήδη υπάρχουσες οδηγίες είναι ξεπερασμένα και για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους επίσης πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστούν αυτά τα θέματα χωρίς νομοθετικά μέτρα. Χρειάζονται νομοθετικά μέτρα, επιγόντως. Συνεπώς, υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες. Η αναπαραγωγική υγεία που πρέπει να προστατευτεί από τους τοξικούς παράγοντες. Πρέπει να προστατευτεί η υγεία από νέους, ε, νέες και το θέμα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πρόγνωση, η αναγνώριση των εργασιακών ασθενειών, αναδυόμενοι κίνδυνοι, από τους οποίους κινδυνεύουν και άντρες και γυναίκες, κάτι το οποίο οδηγεί σε ψυχοκοινωνικούς κινδύνους με αρνητικά αποτελέσματα. Εμείς τον Απρίλιο που μας πέρασε ζητήσαμε νομοθετική ρύθμιση για τις 50 χημικές ουσίες που έχουν κρεθεί ως περισσότερο καρκινογενείς. Η σχετική οδηγία πρέπει να συμπεριλάβει και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Και πρέπει να υπάρξει δράση προκειμένου οι εργοδότες να προστατεύουν τους εργοζόμενους από τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που είναι κυρίως το στρες. Η έρευνα τώρα που έγινε από την υπηρεσία στο Μπιλμπάο στηρίζει όχι μόνο το περιεχόμενο του στρατηγικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις δικές μας εκκλήσεις και απαιτήσει που διατυπώθηκαν στο ψήφισμά μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, λέει πρόεδρος. Έχουμε 30 λεπτά στη διάθεσή μας και δεν έχουμε χρόνο, δεν είχαμε χρόνο να συζητήσουμε αυτό το θέμα το οποίο σαφώς είναι στην κορυφή των προτεραιότητων μας. Το θέμα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, το οποίο και συζητάμε σε διάφορες περιστάσεις. Έγινε η συζήτηση στην Επιτροπή και έχουμε κι άλλο ένα θέμα το οποίο παραμένει στην ημερήσια διάταξη για την Ευρωπαϊκό Έτος στην Ενεργό Γύρανση και για την αλλαγή μεταξύ των γενεών. Έχουμε χρόνο. Μετά τις 6.30 δεν υπάρχει διαρμηνία μπορούμε να πούμε ότι δεν θα γίνει συζήτηση στην Επιτροπή το θέμα αυτό που έχουμε στην ατέντα αυτή τη στιγμή και να περάσουμε κατευθείαν στο επόμενο θέμα και να προσπαθήσουμε να το εκτελέσουμε σε μισή ώρα ή μπορούμε να αναβάλουμε το θέμα για το ευρωπαϊκό έτος για τη γύρανση. Είναι δυνατόν να το αναβάλουμε σε μία μερατική... Όχι. Όχι, λέει ο Πρόεδρος, δεν υπάρχει αυτή τη δυνατότητα. Let's try to really... Ας προσπαθήσουμε να δείξουμε πειθαρχία. And be very short in what we Και να είμαστε πάρα πολύ σύντομοι εφ' εξής. Για να ολοκληρώσουμε και τα δύο σημεία στην ημερήσια καταξία. να ακούσουμε τους κοιόδες εισηγητές για την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστούμε κυρία Κέμπα και ταυτέτε εσείς που βρεθήκαμε στην κατάσταση αυτή να δώσουμε ένα λεπτό το λόγο στον κύριο Μπαχ. Σας ευχαριστώ. Σε 64 λεπτά, λοιπόν θα προλάβω. Νομίζω ότι δεν θα ήταν ευγενικό ε, εναντί των προσκεκλημένων μας να μην κάνουμε τη συζήτηση αυτή. γιατί εκτιμούμε ιδιαίτερα την εργασία τους και νομίζω ότι έθεσαν τα σωστά ερωτήματα και μας έδωσαν τα σωστά κίνητρα. Για μας λοιπόν, για την ομάδα μου, είναι το εξής πάρα πολύ σημαντικό, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά το θέμα του τι κάνουμε με το θέμα των επιπρόσθετων υποχρεωτικών νομικών διατάξεων ο πρόσωπο της ε, Όσερ μίλησε για το, τι δίνει κίνητρο στις εταιρείε. Η νομοθεσία και τα πρόστιμα κατά δεύτερον. Νομίζω ότι από την Business Europe η παρουσίαση είναι λίγο διαφορετική και αυτό μας ε, οδηγεί σε ένα δίλημα. Θα προβούμε σε επιπρόσθετη νομοθεσία ή θα τα αφήσουμε τα πράγματα όσα έχουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μένα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Η κυρία Μάκιντάιερ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν υπάρχει χρόνος να πούμε όσα χρειάζεται να πούμε για την έκθεση αυτή σε ένα λεπτό. Είναι γελίο να το περιμένουμε αυτό. Εγώ θα προτιμούσα πολύ να αφιερώσουμε τη μισή ώρα που έχουμε στο θέμα αυτό και ύστερα να βάλουμε την άλλη συζήτηση. Μια και δεν το κάνετε όμως αυτό, να ευχαριστήσω τον κύριο Κασίνσκι για τη δουλειά που έκανε και να ευχαριστήσω και τους ε, εκπρόσωπους των διαφόρων υπηρεσιών σήμερα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Πολλά φορέζω από την έκθεση αυτή και να πω ότι μου αρέσει ιδιαίτερα το πλαίσιο στην παραγραφό 1, όπου τονίσατε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα σε υψηλού επίπεδου προστασία. Αυτό είναι το σημείο κίνησης, θεωρώ. Θέλω να ρεθεί υπόψη η θέση μικρό μικροεπιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και χαίρομαι που προωθούμε την, ε, τις βέλτιστες πρακτικές. Αλλά θα πρέπει να δείξουμε και μεγάλη προσοχή σε διάφορους τομείς για τους αυθαίρετους στόχους, για παράδειγμα που δεν παίρνουν υπόψη του τι συμβαίνει στα κρατημέλη. Σε κάποιε τομείς λοιπόν θα υποβάλλω τροπολογίες, ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια θετική έκθεση τελικά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βέμπερ, ευχαριστώ τους εισηγητές και τους φιλοξενούμενους τους οποίους ακούσαμε. Τηλεγραφικά να πω ότι είναι σαφές ότι η ασφάλεια στον χώρο εργασίας είναι δικαίωμα αλλά είναι και στόχος. Ένας από τους στόχους είναι να έχουμε μια σωστή οικονομική δραστηριότητα που να επιτρέπει αυτά τα μέτρα ασφαλείας και δεύτερον επίσης να βοηθήσουμε τους εργαζομένους να περάσουν στην τρίτη ηλικία με υγεία. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να αξιολογήσουμε σωστά το τι ισχύει μέχρι τώρα και ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει καλύτερη νομοθεσία, όχι μόνο πιο διαφανής και όχι μόνο στα λόγια, αλλά στις πράξεις. Κάτι το οποίο να είναι κατανοητό από μια μικρομεσαία επιχείρηση που δεν μπορεί να χρησιμοποιεί στρατιές δικηγόρων για να είναι εντάξει. Θα συμφωνήσω επίσης και σε αρκετά από τα θέματα τα οποία έθεσε ο εκπρόσωπος του Business Europe σε σχέση με τους ποσοτικούς στόχους. Οι τροπολογίες λοιπόν, τις οποίες θα καταφέσω και θα συζητήσουμε αύριο, θα έχουν αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Σιλικιώτης. Εγώ θα είμαι πολύ τηλεγραφικός. Πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω με τον εισηγητή, αλλά και τους φιλοξενούμενους. Ε, με αφορμή την κρίση, η εργασία απορριθμίζεται, ε, μεγιστοποιώντας τους κινδύνους που ελοχεύει αυτή η απορρίθμιση με περικοπές στον έλεγχο και την ε, αδυναμία βεβαίω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ενημερώνονται και να κατακτήσουν τι εκτιμήσει κινδύνου σε εργασία. να Ακούσαμε και από τι συζητήσει τέτοια θέματα. Ειδικότερα θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή σε φαινόμενα που φαίνονται σε αυξημένα σε εταιρείε που χρησιμοποιούν υπερεργολάβου ή και τι νέε μορφέ εργασία, όπω παραδείγματο χάρη η εργασία στο σπίτι. Για μα, του αριστερά, είναι σημαντικό το κράτο να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ελέγχου και κανονιστικών ε, πλαισίου για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Το δεύτερο, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι μέρος του συζήτησης με του εργολάβους και την ίδια ώρα να δοθούν τα κατάλληλα εφόδια σε επιτροπέ των εργαζομένων οι οποίε να φροντίζουν για την ενέργεια και την ασφάλεια. Και τελευταίο σημαντικό που τέθηκε από του ομιλητέ, πρέπει να στηρίξουμε τι μικρομεσαίε και τι πολύ μικρέ επιχειρήσει, οι οποίε δεν έχουν τι δυνατότητε να διαμορφώσουν συνθήκε για ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ε, η κυρία Ντέλη. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή και όλους όσοι πήραν το λόγο. Εγώ κρατάω ότι η Business Europe είπε το εξή ότι πρέπει πρώτα να αξιολογήσουμε και μετά να νομοθετήσουμε. Το Δεκέμβριο του 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία τη δικιά μου έκθεση, η οποία ακριβώ αξιολογούσε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Οπότε εμεί την κάναμε αυτή την αξιολόγηση. Και η έκθεσή μου τότε υπογράμμιζε την ανησυχητική κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία που με υποδέχτηκε πολλές φορές στον Μπιλμπάο. Συνεργαστήκαμε συντονισμένα για να υπενθυμίζουμε στοιχεία. Κάθε 5 δευτερόλεπτα έχουμε ένα ε, εργατικό ατύχημα στην Ευρώπη. Αυτό όλοι πρέπει να το έχουμε υπόψη 168.000 θάνατοι. Γιατί δεν νομοθετούμε. 4% του ΕΠ μας. Ε, ναι, φυσικά και πρέπει να δράσουμε. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή και θα συνεισφέρω με πολυάριθμες τροπολογίες. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε. Τέσσερα χρόνια είχαμε σιωπή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μπορεί να έχουμε τέσσερα χρόνια σιωπή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε κυρία Άγκη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Υπάρχουν σημεία στα οποία συμφωνούμε και δεν θα αναφερθώ σε αυτά, αλλά υπάρχουν και κάποιες διαφορές σχετικά με τα δεδομένα τα οποία μας παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν γύρω στις 20.000 επιθεωρητές εργασίας, ένας ανά 9.000 εργαζομένους, 1,5 εκατομμύριο ελέγχων κατέτους. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος εργάζεται 365 μέρες το χρόνο ε, θα υποστεί επιθεώρηση μία φορά ανά 24 χρόνια. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτά θα πρέπει να τα ξαναδούμε για να βρούμε μια άλλη λύση. Τώρα, σχετικά με τις οδηγίες, θα πρέπει οι οδηγίες να είναι πιο απλές, να μειωθεί επίσης και το κόστος των ελέγχων. Ξέρετε ότι η οικονομική κρίση έχει κατασφάξει τις μικροεπιχειρήσεις οι οποίες έχουν τεράστιες δυσκολίες για να καλύψει το κόστος προστασίας των εργαζομένων. Ε, μια καλύτερη χρήση εδώ του κοινωνικού ταμείου μπορεί να δώσει κίνητρα στις μικροεπιχειρήσεις και ένα πλαίσιο νομοθετικό πιο αρμονικό για τους εργαζομένους. Thank Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κύριε Σον Simon. Σας ευχαριστώ. Σε ένα λεπτό. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την ε, Ιουγιουόσα για την ε, μελέτη αυτή που αποτελεί πραγματικά αξιοθαύμαστο έργο και ίσως θα μπορούσαμε σε μελλοντική βάση να στηρίξουμε τις πολιτικές μας σε αυτές τις πραγματικές πληροφορίες. Κατά δεύτερον, δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι συγχαίρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το στρατηγικό πλαίσιο και δεν έχω κάτι προσωπικό κατά, το, κατά των ατόμων που εργάστηκαν, αλλά δεν περιλαμβάνει τίποτα το χρήσιμο. Ε, θα συγχαίρω, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιο θα ήταν το περιεχόμενο. Τέλος, τα τοξικά φάρμακα. Το ανέφερε ένα συνάδελφος ότι πρόκειται για ένα μεγάλο ζήτημα στην ε, ε, υγεία της Ευρώπης. Τα καρκινογόνα φάρμακα που προκαλούν σοβαρές ασθένειες με συστηματικό τρόπο και αυτό το κατανοούν όλοι τα, όλα τα εμπλεκόμενοι φορείς, αλλά δεν αντιμετωπίζεται συστηματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε σε εθνικό επίπεδο και θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί και στα δύο επίπεδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας, λέει Πρόεδρος. Και η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών για την έκθεση αυτή είναι η 30 Ιουνίου το απόγευμα. Όπως σας είπαμε και προηγουμένως όμως, ε, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα ζητήματα αυτά για την ε, υγεία και την ασφάλεια στην μεταργασία αποτελούν βασικό θέμα που απασχολεί την Επιτροπή αυτή και θα εγκρίνουμε λοιπόν την έκθεση σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 23 ε, Σεπτεμβρίου και θα συζητήσω με τη γραμματεία κατά πόσον ε, υπάρχει κάποια δυνατότητα να γίνει μια συζήτηση εις βάθος για το θέμα αυτό. Μια ώρα δηλαδή σε συνεδρίαση της Επιτροπής μετά το καλοκαίρι. Δεν ε, έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν τις συζητήσεις. Θα τις συνεχίσουμε ενδεχομένω μετά το καλοκαίρι. Να σας ευχαριστήσω όλους για το γεγονός ότι ήλθατε εδώ από πλευρά της EU όσα και τον όλα να ευχαριστήσω για το έργο που έκανε παρά το γεγονός ότι ε, βρισκόμαστε σε μια χρονική πίεση κάποια σήμερα. Θα ήθελα να ξέρετε ότι πραγματικά μας έχει εντυπωσιάσει το έργο σας και σίγουρα θα επανέλθουμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή σας αυτή. Και περνάμε τώρα στο 13 της μέρης της διάταξης έχουμε τον κύριο Κούκαν, τον εισηγητή μας, ε, που παίρνει και το λόγο πάρα αυτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω στην παρουσίαση του θέματος, να ξεκινήσω λέγοντας ότι η έκθεση για την εφαρμογή τα αποτελέσματα των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Έτους για την ενεργό και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενναιών ε, προκάλεσε μεγάλο σειρά 184 ε, συγκεκριμένα τροπολογίες. Και αυτό νομίζω ότι καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Και αυτό το καλωσορίζω. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί, θα λάβει η χώρα συνάντηση με τους κοιόντες την επόμενη εβδομάδα, 1η Ιουλίου και ως εκ τούτου είμαι στη διαδικασία προετοιμασίας συμβιβαστικών τροπολογιών όπου αυτό χρειάζεται και γι' αυτό με μεγάλη προσοχή θα ακούσω αυτά που θα μας πούν οι συνάδελφοι και οι σκιώδες από την Επιτροπή για τις τροπολογίες προκειμένου να αποτυπωθούν όλα αυτά στις συμβασικές τροπολογίες τις οποίες και προετοιμάζουν. Για να ξεκαθαρίσω το εξή. θα λάβω υπόψη όλες τις επικοδοματικές ε, παρατηρήσεις εκτός από εκείνες που είναι αντίθετες με την ιδέα της ενεργού γύρανσης ε, και ενδεχομένως ε, όσες ε, ενδεχομένως αποσκοπούν στο να περάσει η συζήτηση σε ένα άλλο επίπεδο. Συνάδελφοι, σε μια τόσο συγκεκριμένη έκθεση αξιολόγησης νομίζω ότι θα πρέπει να επιδραστούμε στα ουσιώδη της έκθεσης και να μην μας πάρει πολύ χρόνο και πολύ προσοχή ένα εντελώς καινούριο στοιχείο. Ο βασικός μου στόχος είναι να παραμείνει συνοπτική και εστιασμένη η έκθεση αυτή για την πραγματική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού έτους 2012 ε, σε ό,τι αφορά την ενεργογύρανση. Πολλές τροπολογίες έγιναν τώρα για την αλληλεγγύη μεταξύ των γενναιών το θέμα αυτό και είμαι γιοτεθειμένος να υποστηρίξω όσες ζητούν μεγαλύτερη έμφαση να δίδεται σε αυτό το τμήμα του 2012. Επίσης θα υποστηρίξω τις τροπολογίες εκείνες που αναφέρονται στις ε, δυνατότητες ε, διαβίου θέση της ανάπτυξης ε, γνώσεων ICT για τους πιο ηλικιωμένους πολίτες και σε ό,τι αφορά τα 50 χρόνια ηλικίας και την συμμετοχή των πολιτών αυτών στην αγορά εργασίας. Επίσης για την καινοτομία. Θα υποστηρίξω τις τροπολογίες αυτές που άπτονται τις καινοτομίες. Δεν θέλω να ξεκινήσω συζήτηση για τις, ε, τα συστήματα συνταξιοδότησης και τη μεταρρύθμιση των συστήματων πρόνοια στα κάτι μελη γιατί πιστεύω ότι αυτό δεν είναι στο πεδίο εφαρμογή τη συζήτηση, αγαπητέ Πρόεδρε. Λοιπόν, προσβλέπω στη συνεργασία με του κοιότε για να προετοιμάσουμε μια καλή έκθεση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο και σκιώδης των σοσιαλδημοκρατών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την έκθεση αυτή. Θα ήθελα όμως να τη συμπληρώσω με κάποιες ιδέες και θα σας τις παρουσιάσω τώρα κάπως σύντομα. Πιστεύω ότι η έκθεση θα πρέπει να υπογραμμίζει ότι η οικονομική και η δημοσιονομική κρίση επιδίνωσε το επίπεδο ένδυας των ε, ηλικιωμένων στην Ευρώπη εξαιτίας ε, του αποκλεισμού των ε, πιο ηλικιωμένων αντιμετωπίσουν δυσκολίες στον τομέα της υγείας και της διατροφής. Υπάρχει και ενεργειακή ένδια. Γι' αυτό λοιπόν δεν μιλάμε μόνο για μία ενεργό ε, τρίτη ηλικία, αλλά και για μια αξιοπρεπή τρίτη εργασία. Θέλουμε λοιπόν να ζητήσουμε από τις χώρες μέλη και τους εταίρους μας να συνεργαστούν για εθνικά πολιτικά προγράμματα που θα διατηρούν στην εργασία ε, τους ανθρώπους μέχρι την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης. Το θέμα δεν είναι να πούμε ότι πρέπει να δουλεύουν πιο πολλοί άνθρωποι μέχρι μια πιο προχωρημένη ηλικία, πρέπει να τους δίνουμε και ό,τι χρειάζονται μέχρι τότε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε ε, τρόπους επίσης να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να δουλεύουν ε, με μερική απασχόληση εφόσον αυτό αποκρίνεται στις ανάγκες τους. Η διαβίου τώρα μάθηση είναι κάτι που πρέπει να υπογραμμίσουμε στα πλαίσια της έκθεσης αυτής. Όσον αφορά τώρα την πρόσβαση στις τεχνολογίες και στην ε, πληροφορική, πρέπει να βελτιωθεί αυτή η πρόσβαση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει μια ψηφιακή στρατηγική που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ενιαίας αγοράς. Έτσι θα βοηθήσουμε τους ηλικιωμένους. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προσωπικά, είμαι υπέρ της διατήρησης του ενεργού βίου στους νέους πρώτα απ' όλα και μετά στους ηλικιωμένους. Πάντως, οι περισσότερες τροπολογίες που διάβασα εγώ νομίζω ότι μπορούν να στηριχτούν. Υπάρχουν πάντως τρεις σημαντικές πτυχές εδώ που θέλω να υπογραμμίσω. Πρώτον, στις τροπολογίες αυτές μιλάμε για τη δημογραφική πτυχή που σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε αυτά στο μέλλον. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς στην Ευρώπη. Να βρούμε τους κατάλληλους πόρους. Δεύτερον, καταρχήν είμαι πολύ επικριτικός στην ε, παράταση του ορίου συνταξιοδότησης και αυτό το active aging δεν νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν άλοθη. Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες των ηλικιωμένων εκτός από την εργασία. Το έχουμε πει αυτό. Υπάρχουν και άλλου είδους, υπάρχει και άλλου είδους συνεισφορά των ηλικιωμένων στην κοινωνία εκτός από την αμοιβόμενη εργασία αυτή καθ' αυτή. Έπειτα, όσον αφορά την τροπολογία 77, είναι μια καλή τροπολογία που θα στηρίξουμε. Εξίσου σημαντικό είναι και το ζήτημα που θέτει η τροπολογία 73 της Άλντε, δηλαδή η προστασία της υγείας. Μπορούμε να αναφέρουμε πολλά παραδείγματα για διακρίσεις που γίνονται σε βάρος των ηλικιωμένων στον τομέα της υγείας, σε πολλές Ευρωπαϊκέ χώρες. Διαπιστώνουμε ότι η πρόσβαση στην υγεία είναι πιο δύσκολη για τους ηλικιωμένου. Πρέπει να το πούμε αυτό και να πούμε ότι υπάρχει διάκριση σε αυτό το τομέα. Κάποια μέρα θα πρέπει να συζητήσουμε και για την ευθανασία. Υπάρχουν και οικονομικές πτυχές, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Η πρόσβαση πάντως την υγεία, το να μην υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος των ηλικιωμένων, εξαιτία της ηλικία δηλαδή, είναι μια πτυχή που πρέπει να υπογραμμιστεί δόντως. Ο Μάικλ από την άλλη Είναι Πολύ καλή έκθεση επιτάπητος και νομίζω ότι έρχεται στη σωστή χρονική συγκυρία. Θα πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν το θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο. Ένα θέμα το οποίο είναι τόσο κρίσιμο για τα κράτη-μέλη, όλα τα κράτη-μέλη μάλιστα. Το θέμα λοιπόν είναι η κατάσταση με τους ηλικιωμένους. Όλοι θα βρεθούμε ηλικία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε ένα σύγχρονο χαρακτήρα στη συζήτηση για του ηλικιωμένου. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα σημαντικά στοιχεία. Δεν θέλω να παρατείνω άσκοπα τη συζήτηση. Η πρόταση τη Άλντερ περιλαμβάνει διάφορε τροπολογίε μαζί με άλλου συναδέλφου εδώ. Και προβλέπω στη συζήτηση με τον κύριο Κούκαν και στη συνεργασία μαζί του να υποδείξω ότι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει μια στρατηγική που θα δώσει απάντηση στο θέμα των δημογραφικών αλλαγών. Παρά τούτου, πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της άνοιας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια ασθένεια που επηρεάζει όλο πιο πολλούς ανθρώπους κάθε μέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βάγκολ. Η κυρία Τσούμπερ έχει το λόγο. Thank you, Chair. Um, uh, quando falamos da implementação deste ano, uh, Ano Europeu do Investimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações, uh, a nossa perspectiva. Uh... Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, καταθέσαμε αρκετές τροπολογίες και στην έκθεση αυτή αλλά και σε προηγούμενες εκθέσεις Και θα πρέπει να πούμε ότι η πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της ε, κάποιων ε, ιδεών γύρω από, την, ε, από τη γύρανση σε σχέση με την συνταξιοδότηση. Δεν θα πρέπει να αναμειγνύουμε αν θέλετε τα θέματα. Νομίζω ότι πολλές φορές η έκθεση επανέρχεται σε αυτού του είδους τις ε, ιδέες. Αντίθετα εμείς νομίζουμε ότι τα δύο αυτά θέματα δεν συνδέονται μεταξύ τους. Νομίζω ότι το θέμα της αύξησης του ορίου ηλικίας είναι ένα από τα κυρίαρχα προβλήματα σήμερα, άπτεται και της παραγωγικότητας τα τελευταία χρόνια Υπάρχουν μελέτες οι οποίες ε, λέγουν, σας θυμίζω, ότι θα πρέπει να μειωθεί ο χρόνος εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας. Και αν λάβουμε επίσης υπόψη μας και τα θέματα γύρω από την ε, βιωσιμότητα της ε, κοινωνικής ασφάλισης, είναι σαφές ότι θα υπάρξει ανάγκη για καλύτερη κατανομή του πλούτου και όχι για παράταση του χρόνου εργασίας. Στις τροπολογίες μας θέτουμε και ορισμένες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές συνδέονται με τον τρόπο με τον οποίο θα ενθαρρυνθεί ο πολίτης να προχωρήσει σε ενέργειες που θα τον βοηθήσουν να περάσει σε μια τρίτη ηλικία με ενέργεια, σε μια ενεργή τρίτη ηλικία με ενεργό τρόπο, όχι με παθητικό τρόπο. Εμείς αυτή τη λογική της οικονομίας της τρίτης ηλικία είναι κάτι το οποίο ε, δεν μας αρέσει, δεν είναι θέμα business ε, η υγεία των πολιτών. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι χωρίς σωστή συνταξιοδοτική κάλυψη δεν υπάρχει περίπτωση να προωθήσουμε την ενεργή γύρανση. Ε, η κυρία Δανούκα, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κούκαν για την έκθεση. Και εμεί καταθέσαμε τροπολογίε. Και νομίζω ότι στη συζήτηση αυτή το βασικό θέμα που συζητιέται και θα συζητηθεί είναι η ηλικία συνταξιοδότηση και η παράδοση του ορίου συνταξιοδότηση. Θεωρούμε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες να εργάζεται κανείς πιο πολύ. Αν αυτό επιλέγει κανείς, γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα επαγγέλματα και οι δυνατότητες απασχόλησης στα διάφορα επαγγέλματα είναι πολύ διαφορετικές. Και θα πρέπει να υποστηρίξει το κράτος τη δυνατότητα αυτή, ως δυνατότητα όμως. Και στις τροπολογίες γίνεται αναφορά στην ε, προσέγγιση βάσει του κύκλου της ζωής, το οποίο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Θα πρέπει να προταθεί σε σχέση με την πρόταση αύξηση του ορίου προσφυγότηση. Αυτέ είναι οι βασικέ προτάσει. Ευχαριστώ πολύ. Η λαγα Άγκερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Παρουσιάσαμε τις τροπολογίες. Ε, γιατί, γιατί έγινε ανταλλαγή μεταξύ των γενναιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και χρειάζεται. Λοιπόν. Πετείται η γυπνίαση των διαφορετικών απόψεων και αυτό θα το πετύχουμε μέσα από τον διάλογο, τον διαφορετικό διάλογο ανάμεσα στους νέους και στους λιγότερους νέους. Και έτσι θα μπορέσει να υπάρξει αμοιβαίος εμπλουτισμός των εμπειριών των μεν και των δε. Ε, θα μπορέσουν να συναντηθούν οι νέοι και οι λιγότερο νέοι και μέσα στους χώρους εργασίας να δημιουργηθεί ένα σωστός διάλογος επικοινωνίας και υψηλής ποιότητας εργασία. Νομίζω ότι σημαντικό είναι και να τονώσουμε ποιοτικά τις ικανότητες της εργασίας των εργαζομένων μέσω της διαβίου κατάρτισης. Η παράδοξη κατάσταση της μακρόχρονης ανεργίας που χτυπά ε, τους ε, νέους από τα 45 και μετά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εκριζωθεί. Τώρα για την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης νομίζω ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι οι κατάλληλες. Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί όταν μιλάμε για την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης. Και αυτό γιατί δεν είναι το ίδιο όλες οι μορφές εργασίας, δεν είναι τόσο κουραστικές όλες. Πρέπει να κάνουμε διακρίσεις και ανάλογα να κρίνουμε. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή ε, πριν να αυξήσουμε το όριο συνταξιοδότησης di, di ottenere comunque un buon documento perché ritengo che comunque eh, la base sulla quale si poggia è estremamente... Νομίζω ότι μόνο τότε θα βρούμε μια σωστή βάση συνεργασίας ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές. Όλους σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Τώρα πρέπει να σας πω ότι στις 15-16 Ιουλίου θα έχουμε το θέμα αυτό. Ε, και συγγνώμη που χρειάστηκε να διαστούμε τόσο πολύ. εφόσον με το λόγο στον κύριο Κούκαν για να συνοψίσει. Ελπίζω να ήταν κάπως εποφελης αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Κύριε Κούκαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο, όχι, ήταν χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν τις απόψεις τους. Κάποιες από τις παρεμβάσεις των σκιωδών εισηγητών, για παράδειγμα των σοσιαλδημοκρατών, θεωρώ ότι αποτελούν μια θετική ε, παρέμβαση για την βελτίωση της ποιότητας του κειμένου και η παρέμβαση του ECR. Να το συζητήσουμε αν θέλετε. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες για τις δημογραφικές εξελίξεις, κάποιες εκ των οποίων είναι πολύ έντονες ως προς τη διατύπωσή τους, νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε μια ρευστική λύση. Μου προκαλεί κάπως έκπληξη. Το γεγονός ότι έγιναν διάφορες παρεμβάσεις και κάποιοι συνάδελφοι έλεγαν ότι ο στόχος της έκθεσης είναι να αυξηθεί το όριο συνταξιοδότησης. Και ότι όλη η συζήτηση εκεί θα εστιαστεί. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Βέβαια το έχω υπόψη μου να αναφέρετε αυτό στην έκθεση και είμαι και κατά. Εξηγήστε μου λοιπόν πώς καταλήξατε στο συμπέρασμα ότι εγώ προτείνω αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, της ηλικίας συνταξιοδότησης. Ευχαριστώ για τις τροπολογίες. Χρήσιμο που κάναμε τη συζήτηση και ξέρουμε λίγο καλύτερα αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε και θα ξεκινήσουν ε, πολιτικές διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρε. Η ευχαριστούμε κύριε Κούκαν. Πολύ γεμάτη η σημερινή συνεδρία Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω όμως ότι πήραμε τις αποφάσεις που έπρεπε να λάβουμε και θα γίνουν και μελλοντικές συνεδριάσεις. Ευχαριστώ πολύ.